Λοιπόν, ξεκινάμε με τις εργασίες της Επιτροπής μας και αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα να χαιρετήσω τον Υπουργό Γεωργίας ε, της Τσεχίας, Γιάκοπ Τσέστα, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου και φυσικά Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας σήμερα με τον Τζάκομπ εξετάζοντας ε, τα όσα μπορείς να ελοπίσει η Τσεχική Προεδρία στο εξάμεινό της και ευθύ αμέσω ε, θα προχωρήσουμε σε συζήτηση η οποία θα μας ε, χρησιμεύσει να συνδέσουμε αυτά τα οποία ο νέος Προεδρεύων Έσκιλ Έρλανσον θα μας ε, αναφέρει σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για το, όπως καταλάβει, τον Υπουργό Γεωργία Σουηδία που ασκεί την Προεδρία. Τζάκομπ, έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου ε, μπροστά από το νέο εκλεγέν Κοινοβούλιο. Είχαμε την Προεδρία του πρώτου εξαμήνου το 2009 και θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και ε, εύχομαι κάθε επιτυχία και στις εργασίες της Επιτροπής σας. Οι σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάντοτε πάρα πολύ καλές, ήταν πάντοτε παραδόσεως καλές και συνεχώς βελτιώνονται. Αυτό είναι ένα, μια πάρα πολύ καλή θετική εξέλιξη διότι ε, μοιραζόμαστε την ευθύνη, για μία από τις πιο σοβαρές, πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η πολιτική αυτή έχει μία τεράστια επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η πολιτική της Γεωργίας. Πιστεύω επίσης ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων θα συνεχιστεί και θα είναι λίαν καρποφόρα στο μέλλον. Έχετε εκλέξει ως πρόεδρό σας ένα πρώην πολύ σημαντικό μέλος του, του Συμβουλίου με μεγάλη εμπειρία ε, των εργασιών του Συμβουλίου και αυτό ε, δείχνει ότι πραγματικά στην εργασία θα είναι λίγα επιτυχής ως πρώην ε, ε, ε, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου θα ήθελα να σας αναφέρω τα συμπεράσματα της Τσεχικής Προεδρίας το, το δεύτερο εξάμεινο του 2008 και το πρώτο εξάμεινο του 2009 υπέφεραν από τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης ε, της διεθνούς ε, αλλά και ευρωπαϊκής. Γι' αυτό η Τσεχική Προεδρία προσπάθησε να βρει έναν ε, συμβιβασμό για την ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική και διέθεσε 5 εκατομμύρια ε, ευρώ για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και αυτή η συμφωνία ε, ε, συγγνώμη πάνω από ένα δις εκατομμύρια ευρώ τα οποία μετακινήθηκαν για το, ειδικά για την ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. αυτή, αυτό το ποσό το διαθέσαμε μετά από τον έλεγχο υγείας, το health check που έγινε πέρσι και επίσης ενισχύσαμε την εισαγωγή του ευ ευρυζωνικού συστήματος ίντερνετ στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ε, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής ανασύστασης συζητήσαμε πολλά εκτακτά προγράμματα ε, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Καν, κανένας τομέας της οικονομίας δεν έμεινε αλόβητος. Ειδικά η γεωργία ε, υπέστη πάρα πολύ, με, πολλές μεγάλες ζημιές και ε, οξύτατα προβλήματα προέκυψαν ιδίως στους παραγωγούς με τη μείωση της ζήτησης του γάλακτος και έτσι ο γαλακτοκομικός τομέας βρίσκεται σε μια εξαιρετική κρίση ε, πρόεδρε, παρακολουθήσαμε πολύ στενά και σε πολύ, με πολύ στενές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξέλιξη και τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα. Πάντοτε ο τομέας του γάλακτος ήταν ε, τομέας προτεραιότητος στις συζητήσεις του Συμβουλίου μας και στις συζητήσεις πάντοτε προσπαθούσαμε να βρούμε μέσα, να βρούμε τρόπους ώστε να αναζωογονήσουμε την αγορά του γάλακτος και να αμβλύνουμε τα προβλήματα των παραγωγών. Και πιστεύω ότι λόγω της κατανόησης της Κομισιόν μπορέσαμε τελικά να κινητοποιήσουμε ε, την στήριξη ε, των εξαγωγικών επιστροφών και των μέτρων ε, αποθήκευσης και την ενίσχυση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη. Επίσης λάβαμε έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα και προτείναμε τα εξής. Μία πρόταση για την επέκταση της περίοδου ε, παρέμβασης, αγορών στην παρέμβαση μετά, πέραν του Αυγούστου φέτος, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η περίοδος του οικονομικού έτους 2010-2011. Ε, ε, παράταση λοιπόν της περίοδου αγορών στην παρέμβαση. Είπαμε ότι η περίοδος ιδιωτικής αποθήκευσης γάλακτος, ε, βουτύρου συγγνώμη, πρέπει επίσης να επεκταθεί με πέραν της 15ης Αυγούστου φέτος. Άλλη πρόταση, πρόταση επιτάχυνσης των άμεσων πληρωμών στους παραγωγούς ε, μέχρι 70%. Ε, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου φέτος. Άλλη πρόταση ε, επίσης, να ενισχύσουμε τους Ευρωπαίους γάλακτου παραγωγούς, πέραν δηλαδή αυτής της γενικής πρότασης, να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα οικονομικής ανασύστασης, που ανέφερα ε, πριν από λίγο. Το Νοέμβριο ε, συνήψαμε μία συμφωνία ε, για την, το health check, τον έλεγχο υγείας της ΚΑΠ. Και έτσι, βάσει της συμφωνίας για τον έλεγχο υγείας, μπορέσαμε να προσαρμόσουμε πολλά μέτρα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τους γαλακτοπαραγωγούς. Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές θα ψηφιστούν από την, στην Επιτροπή σας ε, στα πλαίσια της διαδικασίας απλούστευσης. Ε, λόγω των ε, μέτρων αυτών μπορέσαμε να φρενάρουμε την φθήνουσα πορεία των τιμών του γάλακτος. Όμως δυστυχώς η φθήνουσα πορεία αυτή δεν ανατράπηκε, απλώς ε, σταμάτησε και δεν ανατράπηκε επειδή γενικώ ε, στην παγκόσμια αγορά επικρατούν πάρα πολύ δυσμενείς συνθήκες. Αυτή είναι μια ε, εξαιρετικά σημαντική πρόκληση με τις υπάρχουσες σημερινές συνθήκες η αγορά δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση αυτή για πάρα πολλούς παραγωγούς. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, υπό την Τσεχική Προεδρία ζήτησε από την Κομισιόν να παρουσιάσει μία λεπτομερή έκθεση για τον γαλακτοκομικό τομέα, όπως επίσης μία πρόταση για μέτρα σταθεροποίησης αυτή η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων που θα συνεχιστούν τώρα υπό την Σουηδική Προεδρία. Ελπίζω ότι ε, αυτή η δέσμη των ε, μέτρων που ισχύουν σήμερα αλλά και των μελλοντικών μέτρων θα δώσει ε, μία διέξοδο στους γαλακτοπαραγωγούς από τη δυσμενή τους θέση παρόλα τα μικρά θετικά μηνύματα που είχαμε πρόσφατα στην αγορά, γενικά είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν, να ξεπεραστεί η κρίση αυτή του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη. Αυτή, αυτό λοιπόν θα, θα είναι το βασικό μας έργο, η βασική μας πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε για πολύ καιρό ακόμα στο μέλλον και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αν θέλουμε να επιτύχουμε. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλα σημαντικά θέματα που είχε η μερίσια διάταξη της Τσεχικής Προεδρίας. Η Τσεχική Προεδρία θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ και γι' αυτό το δώσαμε προτεραιότητα στα βασικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας εφαρμογής της πολιτικής. Δηλαδή άμεσες καταβολές στους παραγωγούς μετά το 2014 και επίσης επειδή η συζήτηση του μελλοντικού σχήματος των, δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020 ε, πλησιάζει, κατά την Προεδρία μας ε, ε, έγιναν πολλές ε, ανοιχτές συζητήσεις, ειλικρινείς συζητήσεις για να καθορίσουμε ποια ακριβώς θέματα θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτή τη χρονική περίοδο της ΚΑΠ. Επίσης, η τα μέλη της Επιτροπής σας έλαβαν ενεργό μέρος της συζητήσεις αυτής για το μέλλον της ΚΑΠ και των ε, άμεσων πληρωμών. Το θέμα αυτό ήταν και στην ατζέντα του άτυπου συμβουλίου ε, που έγινε στον Πρνό τον Ιούνιο. Ε, άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας. Η Προεδρία συνεπώς προώθησε προέβαλε μάλλον προ, ε, για το Συμβούλιο του Ιουνίου συμπεράσματα, συμπεράσματα παρουσίασε, τα οποία υποστήριξαν 21 κράτη-μέλη. Η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών έδωσε ένα ε, ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι καταβολές στο μέλλον, οι άμεσες πληρωμές δηλαδή, θα πρέπει να είναι δίκαιες, ε, εύχριστες και λογικές, δηλαδή να, μπορεί, να μπορούμε να τις ε, υπερασπίσουμε σε, ε, σε, σε περίπτωση επικρίσεων. Την ε, συνέχιση του θέματος αυτού θα την αναλάβει η Σουηδική Προεδρία και έχει άμεση σχέση με τον δεύτερο πυλώνα. Τα θέματα του δεύτερου πυλώνα. Η Σουηδική Προεδρία, η Τσεχική Προεδρία επίσης έκανε σημαντικά βήματα πρόοδου για την απλοποίηση ε, των διαδικασιών της ΚΑΠ σε δύο τομείς. Πρώτον, με την ολοκλήρωση ε, του ε, ευρύτατου εινοποιητικού τομέα και ολοκληρώσαμε ένα, μια, την μακροχρόνια διαδικασία πλούστευσης της ΚΑΠ σε αυτό τον τομέα πάνω από 20 κανονισμούς για την κοινή οργάνωση της αγοράς ε, είχαν συζητηθεί επί 12 μήνες, επί ένα χρόνο και συνδυάστηκαν, συγκεράστηκαν σε έναν κανονισμό μέσα στα πλαίσια της απλούστευσης. Δεύτερον, στο Συμβούλιο του Μαΐου, στο Συμβούλιο Γεωργίας και ελήφθη ομόφωνα μια πολιτική απόφαση, έγινε μια πολιτική συμφωνία για το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου επί της απλουστευμένης ΚΑΠ. Το βασικό μήνυμα του Συμβουλίου τότε ήταν ότι η διαδικασία της απλούστευσης της ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχιστεί να, να θεωρείται ως θέμα προτεραιότητος στις τρέχουσες και μελλοντικές συζητήσεις για την ΚΑΠ και το Συμβούλιο επανέλαβε την δέσμευσή του να μειώσει το διοικητικό άχθος κατά 25% μέχρι το έτος 2012 είναι μια πολύ, ένας πολύ σημαντικός συμβιβασμό αυτός που έχει ως στόχο να καταλήξει σε πραγματικά ρεαλιστικά πρακτικά οφέλη ωφέλη για τους παραγωγούς ε, σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής της ΚΑΠ. Κατά την συζήτηση, τις συζητήσεις που έγιναν, τα κράτη-μέλη παρουσίασαν διάφορες ε, συστάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την απλούστευση, όλη τη διαδικασία απλοποίησης της ΚΑΠ και τις εξετάσαμε, τις μελετήσαμε με την πρόθεση να διευκολύνουμε την περαιτέρω συζήτηση και την ανάλυση των προτάσεων αυτών που ε, θα γίνει το Νοέμβριο του 2009 στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα ε, τις συστάσεις των υπηρεσιών πληρωμής των, άμεσων καταβολών. Συνεργαστήκαμε με όλες τις σχετικές διευθύνσεις της Κομισιόν και χρησιμοποίησαμε όλα τα, ε, και συμφωνήσαμε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα της τεχνολογίας για την απλοποίηση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους. Εν συνεχεία επανέρχομαι σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά κατανα... και τους καταναλωτές και τον αγροτικό τομέα και είναι η πολιτική ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα πολιτική ποιότητας. Στο Συμβούλιο του Ιουνίου η Προεδρία της Τσεχίας ε, πέτυχε την ομόφωνη υποστήριξη όλων των κρατών μελών για τα, συμβου... για συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το μελλοντικό μοντέλο του, ε, της ποιότητος, της πολιτικής ποιότητος της γεωργίας και της ποιότητας των τροφίμων και η Κομισιόν εξέδωσε μια ανακοίνωση τον Μάιο του 2009 για αυτό το θέμα. Το σαφές ε, μήνυμα προς τους παραγωγούς είναι το εξής. Θα συνεχίζουμε να τονίζουμε τη σημασία της, πολιτικής ποιότητος και ότι ε, αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των τροφίμων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικά τα έγγραφα αυτά, η ανακοίνωση και τα συμπεράσματα και δείχνουν ξεκάθαρα ότι μας ενδιαφέρει η περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της ποιοτικής ε, πολιτικής για τους καταναλωτές και τα τρόφιμα. Καταρχάς για, την, ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης των προϊόντων, βεβαίως, ε, και για όλες τις συναφείς πτυχές της πολιτικής ποιότητας. Τα ωφέλη της ε, συμφωνίας αυτής είναι ότι δεσμεύτηκαν ε, τα κράτη-μέλη για την, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και επίσης την υποχρεωτική ετικετοποίηση των αγροτικών προϊόντων και μέσα στα πλαίσια της ε, απλούς των διαδικασιών απλοποίησης θα βελτιώσουμε την ετικετοποίηση αλλά και τις ενδείξεις προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης για ειδικά προϊόντα που προστατεύονται. Επίσης είχαμε, η συμφωνία περιλαμβάνει την προστασία ε, ενδείξεων γεωγραφικής προέλευσης από προϊόντα τρίτων χωρών. Η Προεδρία της Τσεχίας ε, διοργάνωσε και μία επιτυχημένη υπουργική ε, διάσκεψη στην Πράγα το Μάρτιο του 2009 με την συμμετοχή αρκετών μελών της Επιτροπής σας. Το αποτέλεσμα αυτής της υπουργικής διάσκεψης συνέβαλε σημαντικά ε, ε, στην επίτευξη συμφωνιών μέσα στο Συμβούλιο υπό την Τσεχική Προεδρία. Παραμένοντας λοιπόν στο, θέματα του πρώτου πυλώνα, ε, θα έρθω τώρα στο θέμα των κανονισμών για το κρέας πουλερικών. Αναλάβαμε την ατζέντα αυτή από τη Γαλλική Προεδρία με, μετά από την ε, καταψήφιση της πρότασης της Κομισιόν για τη, η οποία ε, πρότεινε την ε, χημική επεξεργασία του κρέατος πουλερικών. Αυτό απερίφθη από το Συμβούλιο η πρόταση αυτή. Ήταν ένα ευαίσθητο θέμα ειδικά για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και λόγω της ισχυρής πίεσης ε, που προήλθε από την υπερατλαντική πλευρά. Ε, καταφέραμε λοιπόν να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό για τις, για τις μόνιμες υγειονομικές προδιαγραφές και η Προεδρία έπρεπε να διευρύνει τις ε, προθεσμίες για τα στάντας, για τα πρότυπα που ισχύουν ε, για το κρέας πουλερικών και αποκλείσαμε ε, το κατεψυγμένο κρέας από την, επέκταση του κανονισμού αυτού. Καταργήσαμε δηλαδή τη συμπερίληψη του κατεψυγμένου κρέατος. Επίσης ε, ε, προσθέσαμε ορισμούς συγκεκριμένους που λείπανε από τον κανονισμό και τώρα η νομοθετική πρόταση είναι στα, ε, βρίσκεται στον ΠΟΕ για σχόλια, για σχολιασμό. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, η Τσεχική Προεδρία συνέβαλε όχι μόνο ε, με το πρόγραμμα οικονομικής ανασύστασης αλλά και με το να καθορίσει συγκεκριμένε περιοχές που έχουν handicaps, συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Ξέρετε ότι ο νέος ορισμός των less favored areas είναι ένα πάρα πολύ καυτό θέμα. Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας ενέκρινε τα συμπεράσματα τα οποία βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου μέσω στην οποία τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να λάβουν ε, στην αρχή του 2010 ειδικά μέτρα ενίσχυσης των περιοχών με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, handicaps και την σύνταξη συγκεκριμένων κριτηρίων και ε, χαρτών που θα διευκολύνουν τον καθορισμό των γεωγραφικών περιοχών και των κριτηρίων έτσι ώστε με ενιαίο και διαφανή τρόπο να μπορούμε να ορίζουμε και να, να ταυτοποιήσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές που ε, ε, εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό μετά το 2014 των Less Favored Areas. Όσον αφορά Τώρα, τον φυτοϊγειονομικό και κτηνιατρικό ε, τομέα, θα αναφέρω καταρχάς ένα σημαντικό ε, συμβιβασμό που πετύχαμε, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Στην αρχή της Προεδρίας μας είπαμε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας ε, στον κτηνιατρικό τομέα είναι η ολοκλήρωση του κανονισμού για την προστασία των ζώων την στιγμή της φαγής, ε, στο σημείο της φαγής. Και καταφέραμε μετά από μία σειρά πολύ περίπλοκων διαπραγματεύσεων να επιτύχουμε αυτό το συμβασμό και η πρότασή μας εγκρίθηκε ομόφωνα στο Συμβούλιο του Ιουνίου για τη Γεωργία και την Αλία. Ο συμβιβασμός που πετύχαμε βασίζεται στις τελευταίες επιστημονικές ε, γνώσεις, ε, στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τις τεχνικές παραμέτρους ε, των, του εξοπλισμού των σφαγίων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το σκότωμα των ζώων και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν την οψιόν να εφαρμόσουν τους πιο τους δικούς τους πιο αυστηρούς κανονισμούς, πάνω δηλαδή από το επίπεδο το οποίο αποφασίσαμε εμείς. Το Δεκέμβριο του 2008 η Κομισιόν παρουσίασε μια, ένα σχέδιο οδηγίας στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Η πρώτη μελέτη του κειμένου αυτού ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τροπολογίες του Κοινοβουλίου που συζητήθηκαν. Και τι θα γίνει τώρα, ε, το μέλλον εξαρτάται από την ε, Σουηδική Προεδρία και είμαι πεπισμένος ε, ότι η πρόταση θα ολοκληρωθεί και θα ναι, θα, θα, θα ολοκληρωθεί ε, μέχρι το τέλος του 2009 με τη συνεργασία σας. Όσον αφορά τώρα την ευζοία των ζώων, θα ήθελα να αναφέρω την υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και την ε, γενική ε, δήλωση για την ευζοία των ζώων που ζητούν από τις τρίτες χώρες να υιοθετήσουν τη δική τους νομοθεσία για την προστασία και την ευζοία των ζώων. Μια παγκόσμια διακήρυξη δηλαδή που ε, ζητήσαμε. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την ευζοία των ζώων είναι το σχέδιο οδηγίας για ε, ε, ζωικά υποπροϊόντα. Ζητήσαμε την απλούστευση της διαδικασίας εδώ για τον ορισμό των προϊόντων αυτών για να είναι πιο κατανοητή και πιο διαφανής και για να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις μονάδες και τις ε, αρμόδιες αρχές επιθεώρησης. Αυτό το επιτύχαμε και λάβαμε και υπόψη όλες τις πτυχές της προστασίας της υγείας και των ανθρώπων και των παραγωγών ε, και των ζώων. Όσον αφορά τώρα τον τομέα των τροφίμων, εκεί η Τσεχική Προεδρία κατάφερε να επιτύχει μια πολιτική συμφωνία σε νέα τρόφιμα, νέα προϊόντα ε, στο Συμβούλιο Υπουργών τον Ιούνιο. Η πρόταση ε, στοχεύει ε, στην διασφάλιση της ασφάλειας στην εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την σωστή λειτουργία της αγοράς τροφίμων. Επίσης διευκρινίσαμε ε, ορισμένες ε, ορισμένους ορισμούς ε, τι σημαίνει όρος νέα τρόφιμα και τεχνολογία τροφίμων. Διευκρίνηση λοιπόν ορισμών. Η πρόταση αυτή θα ε, έχει, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για τη δεύτερη ανάγνωση, η πρόταση αυτή. Στην ατζέντα των τροφίμων που συζητήσαμε από την Τσεχική Προεδρία ανήκει και η πρόταση για, έναν, για τον ε, κανονισμό της ε, ετικετοποίησης τροφίμων έτσι ώστε οι ετικέτες να είναι ε, πιο αναγνώσιμες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε Ε, να εξυγχρονίσουμε περισσότερο, μάλλον ε, τις διάφορες πτυχές της, ετικ... ετικετοποίησης, δηλαδή τι συστατικά θρεπτικά περιέχουν και γενικώ ε, το περιεχόμενο των πληροφοριών της ετικέτας. Όλα αυτά παρουσιάζονται, αναφέρονται στην έκθεση προόδου της Τσεχικής Προεδρίας. Και λίγα λόγια τώρα για την, τον φυτοϊγειονομικό τομέα. Η Τσεχική Προεδρία σε συνεργασία με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε έναν συμβιβασμό για τα ε, ζανιοκτώνα ε, και εκεί αντιμετωπίσαμε πολλές διαδικαστικές δυσκολίες και λόγω αυτού η πρόταση ε, δεν έχει ακόμα εγκριθεί, αναμένεται η έγκρισή της και για τα παρασιτοκτόνα και πιστεύω ότι θα εγκριθεί πολύ σύντομα. Και μια άλλη επιτυχία του Συμβουλίου ήταν η έγκριση τριών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των φυτών. Η Τσεχική Προεδρία κατέβαλε προσπάθεια για τον ορισμό νέων διεθνών προτύπων και κριτηρίων του φυτοϊγειονομικού τομέα με στόχο να σταματήσουμε, να εμποδίσουμε τον πολλαπλασιασμό ασθενειών που μεταδίδονται από συσκευασίες που περιέχουν ξύλο. Βάσει του κοινωτικού κεκτομένου συντάξαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία κάλυπταν ορισμένες, ε, ορισμένους πεπαλαιωμένους και μη επιτρεπτούς πλέον τρόπους συσκευασία με συγκεκριμένα υλικά. Ε, επίσης το Συμβούλιο συζήτησε μία πρόταση που περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό για το καθήκον ε, των επιχειρήσεων, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο ξυλίας και ξύλινων προϊόντων. Η Τσεχική Προεδρία προσπάθησε να επιτύχει πρόοδο σε αυτό τον τομέα και καταβάλαμε κάθε προσπάθεια Όμως ε, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και έτσι η πρόταση αυτή θα ζητηθεί περαιτέρω ε, στη Σουηδική Προεδρία. Για τα, τα διεθνή όργανα τώρα τα, τα, και τους διεθνείς οργανισμούς εμείς διοργανώσαμε δύο εκδηλώσεις για την προστασία και την πρόθεση της δασοπονίας τη 19η συνεδρίαση της Επιτροπής Δασοπονίας του ΦΑΟ στη Ρώμη το Μάιο, το Μάρτιο, συγγνώμη, και όπου το κύριο θέμα που συζητήθηκε ήταν η αηφόρος ανάπτυξης, η αλλαγή του κλίματος και η προσαρμογή των πολιτικών της δασ... δασοκομείας ε, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσει. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν, αλλά θα θέλαμε να είχε δοθεί περισσότερη προσοχή ε, στις, στους υπάρχοντες ε, γενετικούς πόρους διεθνώς. Επίσης, ε, συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 5ου Φόρουμ ε, για τα δάση ε, στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα, το Νοέμβριο έγινε αυτό, Νοέμβριο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Α, και τα συμπεράσματα του 5ου αυτού φόρουμ που έγινε τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη τα, τα παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο, συμπεράσματα του Συμβουλίου και κάλυπταν θέματα όπως η προστασία των δασών και του δασικού περιβάλλοντος και την απόφαση ε, του ε, του δημοσιονομικού πλαισίου για την προστασία ε, των δασών και της δασοκομείας. Παρουσιάσαμε και ένα νέο κανονισμό για την προστασία των δασών στο νέο περιβάλλον Αλλά ο κανονισμός για την χρηματοδότηση αηφόρων μέτρων δασοπονίας δεν μπόρεσε να υιοθετηθεί. Επειδή υπήρχαν διαφορές μεταξύ εκείνων των παροχαίων και των, των ωφελουμένων των οικονομικών παροχών. Δηλαδή αυτοί που έδιναν τα κονδύλια της πιστώσης και αυτοί που τελάμβαναν δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Και πιστεύω ότι το θέμα αυτό της χρηματοδότησης, ε, της αηφόρου ανάπτυξης ε, της δασοκομείας ε, θα συνεχιστεί η συζήτηση που τη Προεδρία και θα αποφασιστεί ο κανονισμός το 2011. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, σας έδωσα μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας ως, όταν ασκήσαμε την Προεδρία του Συμβουλίου το πρώτο εξάμεινο και αναγνωρίζω πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει το σώμα ε, σας και ειδικά η Επιτροπή Γεωργίας. Θα πρέπει στην επόμενη περίοδο που θα διανύσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και προκλήσεις που θα πρέπει να λυθούν με κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ε, μια βασική παράμετρο της συνεργασίας μας θα είναι η ικανότητά μας να, να δράσουμε. Η το αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον ε, στο οποίο είναι εκτεθειμένη η παραγωγή μας ε, καθιστά την προστασία του τομέα εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί ενέργειες και γρήγορες ε, αντιδράσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις μόνο ε, με την, μέσω του συνεχούς και εντατικού διαλόγου και της συνεργασίας μας και με την ε, συνεχή βούληση, την πολιτική μας βούληση για συμβιβασμούς και ε, αμοιβαία υποχωρήσεις. Είμαι πολύ ευτυχής που η Γεωργία, τώρα το μέσο της Γεωργίας εμπίπτει στο πλαίσιο της συναπόφασης. Τα ε, μελλοντικά θέματα θα, θα αναφερθούν ε, οπωσδήποτε σήμερα από τον Σουηδό ομόλογό μου και δεδομένου ότι η Σουηδία κατέχει την Προεδρία σήμερα, ε, αυτό το εξάμεινο και οι πολίτες μας έχουν πραγματικά μεγάλες προσδοκίες από μας. Πιστεύω ότι μια καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων είναι και το κλειδί για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και επίλυση και αντιμετώπιση των προκλήσεων. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου εκτίμηση για τη συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας ευχηθώ μια επιτυχή και καρποφόρο συνεργασία στο μέλλον. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Ιακώβε. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία που κάνατε ως Προεδρέμον του Συμβουλίου. Είχατε εξαιρετικά αποτελέσματα ως Προεδρία και είναι βέβαιος πως η Σουηδική Προεδρία θα ακολουθήσει στον δρόμο που χαράξατε. Έχουμε τώρα κάποιες παρεμβάσεις. Ο Άλμπερτ Ντες έχει στήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε από το Συμβουλίο... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για τα όσα έπραξε η Τσεχική Προεδρία. Εγώ προέρχομαι από μια γειτονική σας περιοχή. Εκλέγομαι σε μια περιφέρεια που γυπνιάζει με την ε, <clears throat> χώρα σας. Πραγματικά οι εργασίες που κάνατε ήταν πολύ Σημαντικέ, αλλά αντιμετωπίσετε κάποιε δυσκολίε λόγω τη ιστορικής πολιτική κατάσταση της χώρα σα. Πάλι συγχαρητήρια για τα όσα μπορέσατε να κάνετε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα τα θέματα που εσείς στήξατε, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Εσείς αναφερθήκατε στο ζήτημα του γάλατος. Το συζητήσαμε το ζήτημα χθε με την κυρία Επίτροπο. Εισαγάγατε κάποια μέτρα αλλά εγώ θα είχα προτιμήσει ε, αντί της παρεμβάσεως να είχαν αυξηθεί οι ενισχύσεις προς το βούτυρο έτσι ώστε οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν να ευνοηθούν και να απορροφήσουν αυτό το αυτές τις ποσότητες ε, διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Μιλήσατε και για το ε, μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής που θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Αναφερθήκατε επίση και στον τρίτο πυλώνα και για τις ε, πλέον μειονεκτούσες περιοχές. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν κύριε Υπουργέ να φροντίσετε μαζί με τους συναδέλφους και με τους ισχύοντες περιορισμούς με αυτές τις, σε αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές που δεν είναι ορεινές περιοχές αλλά παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα για λόγους κλιματολογικούς ε, και άλλους. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να φροντίσετε να παραμείνουν σε αυτήν την κατηγορία διαφορετικά θα μπορούσαν να διατηρήσουν την, γεωργία την γεωργική τους παραγωγής. Αναφερθήκατε και στην ποιότητα της παραγωγής Γνωρίζουμε πως ε, στην Ευρώπη έχουμε πολύ υψηλά στάνταρ ποιότητας. Πρόβλημά μας είναι πως ε, αυτή η υψηλή ποιότητα δεν ε, ανταμείβεται επαρκώς θα λέγαμε την αγορά. Δεν, πληρώνουμε, δεν υπάρχει σωστή σχέση ποιότητας κόστους. Αναφέρομαι στα γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας Έχουμε επίσης και εξαιρετικά κρασιά και η αμπελοπαραγωγή και θα πρέπει να δεν ανταμείβονται ικανοποιητικά. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και να εφαρμόσουμε μια καταλληλότερη πολιτική. Επιθύνω λοιπόν σε εσά, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να φροντίσετε να τηρούνται τα πρότυπα τα δικά μας και στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ε, ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής γεωργίας. Τώρα, σε ό,τι φορά τα πουλερικά, σε είμαι που εσείς ε, δεν υπαναχωρήσατε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια σε επίπεδο παραγωγής τα παραγωγικά πρότυπα θα πρέπει να τηρηθούν από όλου ε, του ε, εταίρους μας από τους οποίους εισάγουν προϊόντα. Επίσης αναφερθήκατε στον ρόλο της ε, Επιτροπής μας, ο οποίος θα αυξηθεί, θα γίνει πιο σημαντικός μέσω της συναπόφασης. Αλλά κύριε Υπουργέ, πότε θα ξεκινήσει αυτή η συναπόφαση, πότε η κυβέρνησή σας η χώρα σας μάλλον θα υπογράψει αυτήν την συνθήκη της Λισαβόνας, ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε πότε η Τσεχία θα συνεισφέρει προκειμένου να καταλήξουμε στην συναπόφαση. Κατά τα υπόλοιπα σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Σε ευχαριστώ, Άλμπερτ. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Χθε, ε, Τζάκοπ, συζητήσαμε αυτό το θέμα της ενιαίας εφαρμογής των ε, προτύπων και των κανόνων ασφαλείας, ε, δίχως να θέλουμε να γίνουμε ή να διολυστήσουμε στον προστατευτισμό. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, τα πρότυπα αυτά να τηρούνται και από όσου εξάγουν στην Ευρώπη. Λουίς Σάντος να κάπως έχει το λόγο. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών θα ήθελα και εγώ να σας χαιρετήσω Μας κάνατε μια παρουσίαση των ε, δραστηριοτήτων της Προεδρίας σας και μας είπατε ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες για την Τσεχία και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όμως πρέπει να πω ότι για μια χώρα που θεωρείται μάλλον ευρωσκεπτιστική. Νομίζω ότι χειριστήκατε τα πράγματα αρκετά καλά και νομίζω ότι καταφέρατε να ανταποκριθείτε στις διάφορες προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ε, σώμα ε, που είναι ε, κοντινότερο στους πολίτες και γνωρίζετε ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το γαλακτοκομικό τομέα η Προεδρία σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν πολλές προσπάθειες, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Πολλές φορές ε, εξετάστηκε το θέμα αυτό από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεδριάση της δικής μας Επιτροπής ε, και από τότε τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανοποιητικέ οι προσπάθειες της Τσεχικής Προεδρίας, αλλά ε, θα ήθελα να γνωρίζω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ε, επίλυση του σοβαρού προβλήματος του γαλακτικομικού τομέα στην Ευρώπη. Grazie Luis. Ευχαριστώ, Λουίς. Κύριο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τα όσα πέτυχε η Τσεχική Προεδρία ήταν η ε, πρώτη προεδρία μιας ε, νέας ε, χώρας, νέας ελθίσας χώρας. Ασχολήθηκατε με ζητήματα πολύ περίπλοκα και πραγματικά είχατε εξαιρετικά αποτελέσματα. Εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στο ζήτημα της πρότασης κανονισμού για την προστασία των ζώων κατά της φαγής. Ήταν συζητήσεις ιδιαίτερα ε, φορτισμένες συναισθηματικά. Ε, γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα, διότι ήμουν εισηγητή ε, από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου. Γνωρίζω λοιπόν καλά ποια ήταν η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έγιναν οι όλες οι συζητήσεις. Ε, σας συγχαίρω λοιπόν για τα αποτελέσματα τα οποία καταλήξατε. Και ελπίζω πως η Σουηδική Προεδρία θα είναι εξίσου αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Δεν έχουν στήσει άλλη το λόγο. Να δώσω το λόγο στον ε, Τζάκομπ ε, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι και τον ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδείτε το λόγο πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω πως ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα πετύχαμε ως τσεχική προεδρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίσανε και ορισμένοι εξημών. Η κατάσταση που επικρατεί στην ε, αγορά του γάλακτος ε, νομίζω πως δεν θα πρέπει να μας ικανοποιεί. Η κατάσταση όμως είναι ιδιαίτερα περίπλοκη όπως γνωρίζουμε. Αυτή η κρίση που πλήττει τον τομέα του γάλακτος είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε εκ του και σίγουρα απαιτούνται περισσότερα μέτρα. Πρέπει να έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της ε, παρέμβασης αλλά και της ε, και της αποθήκευσης αν θέλετε των προϊόντων αυτών. Χρειάζεται ως εκ τούτου να δραστηριοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ως εκ τούτου εγώ εξετίμησα ιδιαίτερα τον ρόλο που έπαιξε και συνεχίζει να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κατάσταση στην αγορά γάλακτος είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε επανειλημμένα και την Κομισιόν αλλά και το Συμβούλιο και θα συνεχίσει να μας απασχολεί στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ε, υπόθηκε ότι πέραν των όσων γίνονται η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κατορθώσαμε να βάλουμε μια τροχοπέδη ε, κρίση και η κατάσταση πιστεύουμε πως σύντομα θα βελτιωθεί. Θα καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες ε, μελλοντικά. Έχουμε μια σειρά προτάσεων και μέτρων που προέρχονται από τους υπουργούς ε, των κρατών μελών που έχουν κάποιες απόψεις έτσι ώστε να μπορέσει ο τομέας ε, να ξεπεράσει την κρίση που αντιμετωπίζει. Poslanec στο θέμα της ε, ποιότητας ε, και των προτύπων. Καταλαβαίνω απόλυτα τις ερωτήσεις αυτές. Εγώ για πάνω από 30 χρόνια έχω ε, εργαστεί για θέματα ασφάλειας και ποιότητας ε, των ε, προϊόντων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είμαι 100% σύμφωνος ότι οι καταναλωτές μας θα πρέπει να αγοράζουν ασφαλή και προϊόντα, και ποιοτικά. Οι, τα, οι κανόνες και τα πρότυπα θα πρέπει να τηρούνται τα τρόφιμα που βρίσκονται στην αγορά θα πρέπει να πληρούν τις ε, προδιαγραφές και αναφέρομαι εδώ ειδικότερα στις εισαγωγές τροφίμων. Ε, δεν μπορούμε εμείς, οι δικοί μας και παραγωγή να τηρούν τα πρότυπα και να μην εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες για τα προϊόντα τα οποία εισάγονται. Επίσης ε, τέθηκε μια ερώτηση για ένα ζήτημα το οποίο έθιξε κάποιος ακροθυγός το συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω πως η συνθήκη της Λισαβόνας θα εγκριθεί, θα κυρωθεί από όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη και θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή στην οποία τόσο προσβλέπουμε. Ωραία. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Τσέχο Υπουργό, ευχαριστώ Τζακόμπ. Ελπίζω ότι από τον Οκτώβριο αυτή η συνεργασία θα γίνει πραγματικότητα. Εμείς πάντως συμπεριφερόμεθα και εργαζόμαστε ως αν ήδη να υπήρχε η συναπόφαση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αποχαιρετήσω τον ε, Υπουργό. Θα, θα προχωρήσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ελπίζω όχι να, όλοι να έχετε τις κάρτες σας. Ένα λεπτό λοιπόν για να αποχαιρετήσουμε τον ε, κύριο Υπουργό και επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας άμεσα. Bene, diamo inizio allora a questa sequenza Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Πρώτο σημείο. Θα πρέπει να ψηφίσουμε με απλοποιημένη διαδικασία το θέμα της παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα στη σκόνη. Όπως είπαμε και σήμερα το πρωί με τους συντονιστές, αλλά και όπως επανειλημμένα τονίστηκε χθε τη παρουσία της ε, Επιτρόπου Μαριάν Φίσουμπολ. Μπολ, όλοι εδώ στην Επιτροπή, ζητάμε να γίνει κάτι παραπάνω. Ο γαλακτοκομικός τομέας βρίσκεται σε βαθιά κρίση και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν και σήμερα το πρωί αναφέραμε την ε, ιδέα να αναγγείλουμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου προτάσεις ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες για το θέμα του γάλακτος, αλλά και δεν αποκλείουμε για μια πρόταση πρωτοβουλία συγκεκριμένη για την κρίση του γαλακτοκομικού τομέα που θα αξιολογήσουμε μετά από το έκτακτο συμβούλιο της προσεχούς Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου και μετά από αυτήν την συζήτηση στην Ολομέλεια, κατά την οποία θα παρουσιάσουμε το αίτημα της προφορικής ερώτησης ε, μετά από σχετικές προτάσεις των ομάδων. Αλλά και χθε, όπως και σήμερα το πρωί στο πλαίσιο των συντονιστών, συμφωνήσαμε την αναγκαιότητα να στείλουμε άμεσα ένα ισχυρό μήνυμα το οποίο θα καταδείξει ότι αυτή η Επιτροπή είναι μια Επιτροπή που θέλει να είναι αποτελεσματική στις επιλογές αλλά και θέλει να το πράξει προτού να τεθεί ακόμα σε ισχύ στην απόφαση που θα συμβεί εάν και όλοι το ευχόμαστε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία έχει αίσιο πέρας. δώσω τον λόγο στον ε, Λουίς ε, θα ήθελα να έχω την βεβαιότητα πως ουδής εξημών με ύψιλον αντιτίθεται στην πρόταση τροπολογίας για μια πρωτοβουλία για τον νομικό τομέα και για το βούτυρο. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που θα αφορά στην αποδίκευση των τυριών εμείς λοιπόν θα αποκαραστήσουμε αυτή την θέμα της αποθήκευσης. Τώρα, ο Λουίς Κάπουλα Σάντος θα μας μιλήσει για αυτή την τροπολογία, θα πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην Κομισιόν αλλά και προς το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν πως όλοι θα συμφωνήσετε όπως συμφώνησαν και σήμερα το πρωί οι συντονιστές σας και να μην αντιταχθείτε σε κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένο να ερωτήσω εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που αντιτίθεται σε αυτήν την διαδικασία. Να δώσω το λόγο στον Λουίς Κάποντα Σάντος. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση μου ουσιαστικά συνεχίζει την ε, απόφαση στην οποία είχαμε καταλήξει και δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να δώσει ένα μήνυμα αλληλεγγύης ε, με το Συμβούλιο, ότι μπορούμε δηλαδή να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο για να ε, αντιμετωπίσουμε την κρίση. Μπορούμε να πούμε επέκταση του μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσης ε, για το ε, τυρί, δηλαδή να υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός που υπάρχει και για το βούτυρο και ελπίζω ότι θα λάβουμε την απαραίτητη στήριξη για την πρόταση αυτή. Σιλβέστη, έχεις το λόγο. Ναι, αν πρόκειται να συζήτηση, βεβαίως, πρόεδρε. Όχι, δεν υπάρχει συζήτηση, άρα όχι. Λοιπόν, αν όλοι συμφωνούμε θα προχωρήσουμε ούτως και σας ερωτώ εάν συμφωνείτε με την τροπολογία. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις. Και αν υπάρχουν και αποχές. Δεν πρόκειται για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή. το χειρός. Λοιπόν, άρα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε. La votazione elettronica non è necessaria. Abbiamo soltanto bisogno... Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία. ψήφι υπέρ της τροπολογίας. Διανατάσεως του ισχυρός. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εγκρίνεται ως νομοθετική τροπολογία. Αφού εγκρίθηκε λοιπόν η τροπολογία, θα πρέπει να εγκρίνουμε και την πρόληψη νομοθετικού περιεχομένου για το γάλα και το βούτυρο. Συμφωνείτε? Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. αποχές. Λοιπόν, ομοφόνος εγκρίναμε να παραταθεί η περίοδος ε, παρέβασης ε, και για το, για το βούτυρο και συμπεριλάβαμε και μια τροπολογία για, την, ε, για να ισχύσουν για το τυρί τα όσα ισχύουν για το βούτυρο σχετικά με την αποθήκευση θα μάθω σιγά σιγά και θα τα κάνω καλύτερα και πιο γρήγορα. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν. τα άμεση στήριξη για του γεωργού στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική. Και εδώ πρόκειται η ψηφοφορία με απλοποιημένη διαδικασία. Ήταν ένα θέμα ιδιαίτερα εθνικού χαρακτήρα, αφορούσε στον προπολογισμό τη διάρκεια τελευταία συνεδριάσεω. Είχαμε αποφασίσει να εφαρμόσουμε την απλοποιημένη διαδικασία για αυτόν τον φάκελο, όπω βλέπετε στο άρθρο 46, παράγραφο 1. Υπάρχουν ενστάσει. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, η έκθεση είναι δεκτή. Και τώρα θα περάσουμε σε μια πιο δύσκολη διαδικασία. Πέραμε στον προπολογισμό, προπολογισμό 2010, τμήμα 3. Προτού να περάσουμε στις οφορίες, θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε on block, ομού, τις τροπολογίες που αποκαθιστούν το προσχέδιο προϋπολογισμού. Με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι οι μόνες τροπολογίες που αφορούν τη συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού. Κυρία Γέγκλε θέλει να λάβει το λόγο που πρέπει στις ψηφοφορίες. Όχι. Ωραία. Λοιπόν. Ε, Εάν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία on block όλων των τροπολογιών που αποκαθιστούν την αρχική γραμμή του προπολογισμού. Εδώ χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πολύ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 33 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, μία αποχή. Δεκτά, δεκτές μάλλον. Και τώρα ψηφίζουμε τις επιμέρους τροπολογίες ενώ έχουμε εγκρίνει τα αρχικά ποσά. Προχωράμε στις ψηφοφορίες λοιπόν. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με το μηχάνημα. Αν δεν λειτουργήσει τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες διανατάσσεως της χειρός. Λοιπόν, περνάμε στις ψηφοφορίες ε, ανατροπολογία. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία διανατάσεως της χειρός, διότι ε, το πρόβλημα είναι τόσο ε, η μηχανή, αλλά και το ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη τροπολογία 52-52. Πενήντα 52, 52 τροπολογία. Ο Λεφόλη ζήτησε τον λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω χωριστή ψηφοφορία ε, επί τη τροπολογία αυτή, διότι υπάρχουν πολλέ ε, υποτροπολογίε που αφορούν ε, διάφορα προϊόντα. Αυτή τη χωριστή ψηφοφορία την θέλουμε επί των δύο πρώτων γραμμών και όλα τα υπόλοιπα on block. Λοιπόν, διαχωρίζουμε τα δύο πρώτα τμήματα της τροπολογίας ή τις δύο πρώτες τροπολογίες από όλες τις υπόλοιπες. Στεφάν, αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα και εγώ να πω. Περνάμε σε χωριστή ψηφοφορία και όχι το σύνδετο της τροπολογίας, αλλά για ορισμένα προϊόντα αρχικά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμεθα στην κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή μόνο για τα δημητριακά. Λοιπόν, κατάργηση των επιστροφών μόνο για τα δημητριακά. Ψήφι Okay. Chi è contrario all'eliminazione delle Ψήφι κατά της κατάργησης ε, των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Bene, e adesso chi si astiene? Αποχές. Bene, è stato rigettato. Απορρίπτεται. Και τώρα στο δεύτερο τμήμα, δηλαδή την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Η 52-52 λοιπόν απορρίφθηκε στο σύνολό τη Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 52-01. 52-01. Τη βρήκατε. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Η 5201 έγινε δεκτή. 52 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 52-71 κατά αποχές τροπολογία απερίφθη τροπολογία 53-27. 53-27. Η ομάδα των Πρασίνων θέλει να λάβει το λόγο. Μάρτιν. Συμφωνούμε ότι θα μπορούσαν τα ποσά αυτά να προέλθουν από την ε, παρέμβαση. Περνάμε. Devo chiedervi se c'è qualcuno contrario. Υπάρχει κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που αντιτίθενται, δεν θα ψηφιστεί. Διαφορετικά μπορούμε να περάσουμε στην ψήφισή του. Πρόκειται για προφορική τροπολογία. Είστε όλοι υπέρ. Λοιπόν, περνάμε στην ψήφισή της. 53-27 θα ψηφιστεί χωρίς αυτά τα όσα ανέφερε ο Μάρτιν. Ψήφι υπέρ. Ψήφι Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην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 52-58. Τροπολογία 52-58. Ψήφι ψηφιπερ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5205. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5319. ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 53-18 ψηφιπερ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5209. Ψήφι κατά αποχές η τροπολογία έγινε δεκτή 52-10 ψήφι κατά εποχές Δεκτή. Τροπολογία 52-75. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. τροπολογία 5260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5281 τροπολογία ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται 52-84 έχει αποσυρθεί. 52-93. 52-93 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές τροπολογία είναι δεκτή. 52-72 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 52-73 Κατά. περ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία έγινε δεκτή. Πού θα πάει θα τελειώσουμε. 52-87. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53-17. Α, όχι, όχι, όχι. Λάθος.

Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5288. Πρόκειται για προφορική τροπολογία των πρασίνων. Πρέπει να συμφωνούμε όλοι. Μάρτιν. Θέλουμε μία συμπλήρωση και θα τη διαβάσω στα αγγλικά. έτσι ώστε να επιτρέψει στο τομέα να αναπτύξει μία αηφόρο σχέση μεταξύ της ε, ε, προσφοράς και ζήτησης. Ψηφίζουμε λοιπόν, όχι, συγγνώμη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Το μικρόφωνο κάνει διακοπές. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Εάν, ε, νομίζω ότι η ομιλήτρια είπε, εάν προσθέσουμε τις ενώσεις παραγωγών και συνεταιρισμού. Αν προσθέσουμε αυτά τα δύο μπορούμε να δεχτούμε τροπολογία. Αλλά δυστυχώ δεν λειτουργεί το μικρόφωνο τη. Η ΣΥΔΙΑ λέει εκτό από τι οργανώσει, τι ενώσει ε, των καταναλωτών αλλά και του συνεταιρισμού ε, των παραγωγών συγγνώμη και του συνεταιρισμού. Εντάξει, με αυτή τη διόρθωση μπορούμε να ψηφίσουμε. 52-88 με αυτή την τροποποίηση επεκτείνοντας το σε όλους. Ψήφι πέρα. Κατά. αποχές. Με 52-88 έγινε δεκτή. Τροπολογία 53-26 το πρώτο τμήμα. 53-26 ψηφιπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται υπήρχε πρόβλημα με την διερμηνία από τα γερμανικά Εντάξει, αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα. 52-89 τροπολογία. Ψηφιπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 52-90. Ψηφιπέρ. κατά εποχές δεκτή 52-16 ψήφι περ κατά αποχές δεκτή 52-51 υπέρ Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Τις 52-51. Κατά. Η τροπολογία έγινε δεκτή. 52-17. Υπέρ. κατά αποχές δεκτή 52-18 υπέρ κατά αποχές δεκτή

contrario? Κατά. Απορρίπτεται. 52-67. Υπέρ. Κατά. αποχές δεκτή 52-55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53-11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52-61 χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της 5261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 52-69 υπέρ κατά αποχές

κατά αποχές δεκτή 53-29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52-91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52-49 ψήφι κατά αποχές δεκτή προπολογια 52 52-62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52-68, 52-68, υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. Πενήντα εβδομήντα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τώρα η τελευταία 52-31 υπέρ Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, έχει συμπεριληφθεί. Άρα, τελειώσαμε. Allora, prima di dare il via Λοιπόν, προτού να περάσουμε στην ε, παρουσίαση της μελέτης αντικτύπου, σας προτείνω το περάσουμε στο τελευταίο σημείο, σημείο 14. Πρέπει να ψηφίσουμε προκειμένου να υπολουθεί ερώτημα με προφορική απάντηση σχετικά με την κρίση που βιώνει ο τομέας του γάλακτος. Συζητήσαμε στο πλαίσιο των συντονιστών σήμερα το πρωί. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να πάμε στην Ορμέλη και να συζητήσουμε το γαλακτοκομικό πρόβλημα. Ζητώ λοιπόν από τους προέδρους, λέει μάλλον τους συντονιστές εννοεί, ε, να ετοιμάσουν λοιπόν την ερώτηση για την Ολομέλη. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα στο πλαίσιο ή μια έκθεση στο πλαίσιο τη Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσω από όλε τι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν ε, ψηφίσματα με την ευκαιρία της ε, Ολομέλειας. Επειδή είναι ιδιαίτερα σοβαρό το ζήτημα, παρακαλώ να προχωρήσουμε ούτω εκτό αν υπάρχουν ενστάσεις δεν υπάρχουν στάσεις. παρακαλώ οι πολιτικοί ομάδε να προετοιμαστούν για την Ολομέλεια του Στρασβούργου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε, μια που ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας, να περάσουμε στο σημείο 13, που πρόκειται για την παρουσίαση μιας μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστου ε, λειτουργίας ε, της κτηνοτροφίας για την παραγωγή κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χαιρετήσω τον κύριο Φιλίπ Κοτό και την ε, κυρία Αν Κοτέ και τους κυρίους Πίτερ Χόρτ και Πίτερ Χόρτ που θα μας παρουσιάσουν την ε, μελέτη σχετικά με ε, τις επιπτώσεις από το αυξανόμενο κόστος της κτηνοτροφίας. Κύριε Κοτό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η μελέτη αυτή ανταποκρίνεται σε αίτημα του Κοινοβουλίου της προηγούμενης Επιτροπής Γεωργίας ε, του Κοινοβουλίου σας και στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναλύσει την κατάσταση μετά από την ε, αύξηση των τιμών της ενέργειας, ε, των ελέγχων σπόρων κλπ. Να αξιολογήσουμε λοιπόν τον αντίκτυπο για το σύστημα παραγωγής κρέατος στην Ευρώπη να εντοπίσουμε τις αδυναμίες ε, στο σύστημα ακτινοτροφίας, ε, να δούμε ποσοτικά τι μέγεθος έχει αυτή η κρίση και πώς μπορεί να εξελιχθεί κατά τα επόμενα έτη και βεβαίως ε, να κάνουμε και κάποιες προτάσεις. Η μέθοδος που επιλέξαμε είναι καταρχάς ε, να επικεντρωθούμε στην περίοδο 2004 2008. Το 2004 το 2006 τα πράγματα ήταν αρκετά σταθερά και μετά το 2007 2008 είναι η περίοδος έκρηξης του λειτουργικού κόστους, ειδικότερα για τους ε, ε, κρεατοπαραγωγούς. Ε, επιλέξαμε επίσης ε, να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένους τύπους. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το ρίκα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα διαθεσιμότητας με το ρίκα για τα δεδομένα 2007 και 2008. Δεδομένου λοιπόν ότι είχαμε λίγα μέσα στη διάθεσή μας, προσπαθήσαμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες χώρες για το βοδινό κρέας Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, για το αρνί ε, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, για το χοιρινό Γερμανία, Γαλλία, κάτω χώρες Πολωνία και για, την, ε, για τα πουλερικά Γαλλία, ε, κάτω χώρες και Πολωνία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα μεθοδολογικό είναι ότι ε, οι υπολογισμοί μας γίνονται σε ευρώ και έτσι δεν συνυπολογίζονται οι διαφορές λόγω των ισοτιμιών, ε, για παράδειγμα του πολωνικού σλότη ε, και της αγγλικής λύρας. επίσης, μιλούμε για πραγματικό κόστος λειτουργίας και ε, μιλάμε για πιο ε, ε, ευκαιριακό κόστος, για συγκυριακό κόστος για τους για την οικογενειακή εργασία και το κεφάλαιο. Πρόκειται για μια δύσκολη μελέτη γιατί αφορά τέσσερις διαφορετικούς τομείς, 11 εμπειρογνώμονε από 8 διαφορετικές ε, οργανώσεις ε, ε, και μάλιστα από 5 χώρες. Είχαμε πολλούς εμπειρογνώμονε από τις κάτω χώρες και από το Ίδρυμα Κτηνοτροφίας που εδρεύει στη Γαλλία. Βλέπετε στη διαφάνεια για την αύξηση των, του κόστους βλέπετε ποια είναι η διαφορά για το κρυθάρι, ε, για τη βρώμη, οι οποίες τιμές παρέμειναν σχετικά σταθερές ε, από το 2004 ως το 2006, άρχισαν να αυξάνονται το 2007 και έφτασαν στην κορύφωσή τους το 2008. Ε, υπήρξαν λοιπόν πολλές περιπτώσεις ε, αύξησης των τιμών ε, κυρίως το 2000 και το 2007 και 2008, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξε αύξηση του κόστου το 2004 έως 2006. Επίση, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τη μελέτη μας με την αύξηση των τιμών ενέργειας. Βλέπετε εδώ στην κορυφή με κόκκινο χρώμα. Βλέπετε ότι αυξήθηκε και η τιμή του πετρελαίου από το 2000 ε, ήδη, μετά το 2004 επιπλέον κλπ. Και υπήρξε μια μάλλον καθυστερημένη ε, επίπτωση στις τιμές ε, στην γεωργία. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι είναι αρκετά εφήμερε οι μεταβολές του κόστους ε, στα γεωργικά προϊόντα και είναι μάλιστα πολύ συγκυριακή αυτή η αύξηση. Τώρα, για το σύστημα παραγωγής του κρέατος. Ποιες είναι οι συνέπειες. Βλέπετε για παράδειγμα το κρέας ε, ε, τις εγκαταστάσεις πάχυνσης βλέπετε πώς ε, είναι η εξέλιξη από τις αρχές του 2000 βλέπετε ότι υπάρχει μια αύξηση, μια κορύφωση το 1985 από το 2000 έως το 2006 υπάρχει μια σταθερότητα και από το 2006 υπάρχει μια πραγματική έκρηξη η οποία είναι τελείως ε, διαφορετική και αντίστροφη με τη μείωση των τελευταίων 10 ε, ετών. Δεν είναι βέβαια η κατάσταση ίδια σε όλες τις χώρες. Βλέπετε για παράδειγμα για την πάχυνση των χείρων ε, στις διάφορες χώρες. Είναι αρκετά σταθερά ε, τα πράγματα, ειδικά για την πάχυνση των χείρων. Όσον αφορά τώρα την τιμή της ενέργειας, βεβαίως έχουν μια άμεση επίπτωση ε, στις, στην κτηνοτροφία. Ειδικότερα, για παράδειγμα, το, οι τιμές του λιπάσματος έχουν άμεση σχέση με την ε, τιμή ε, των ε, με την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου. Απλώς υπήρξε δεν υπήρξε σταθερότητα, δεν υπήρξε μείωση παράλληλα με την, μείωση, με την, αύξηση των, με, την, με τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Με την, με το παράδειγμα, με το παράδειγμα κυρίως να αφορά το 2008 και 2009. Επίσης, ε, στη συνέχεια ο συνάδελφος θα σας ε, μιλήσει για ε, το χοιρινό και τα πουλερικά. Εγώ θα μιλήσω για το βοδινό και το αρνίσιο κρέας. Βλέπουμε για παράδειγμα τι γίνεται στην κατάσταση, με την κατάσταση ε, βοδινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπλοκα τα πράγματα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με άλλες περιοχές στον κόσμο, γιατί είναι δύο τρίτα, ε, δύο τρίτα των αγελάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι γαλακτοφόρες. Επομένως, Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της κατάστασης του ε, ε, βοδινού κρέατος και ε, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του, γαλακτικού τομέα, του γαλακτοκομικού τομέα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν, οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε μία μικρή διάκριση μεταξύ των εκμεταλλεύσεων βοδινού κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται και στα δύο. Το διάγραμμα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά έχετε και την ε, ε, γενικότερη έκθεση όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που δείχνει είναι ότι διαφορετικό το κόστος της παραγωγής ε, στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες ασχοληθήκαμε από 3,30 από ανασφάγιο μέχρι 4,80 ανάλογα με το είδος συστήματος που εφαρμόζεται. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες διαφορές. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και τεράστιες διαφορές ε, στη σύνθεση του κόστους παραγωγής. Ε, βλέπετε για παράδειγμα διαφορά 8 έως 25% για το κόστος ε, των τροφίμων. Και κάτι ακόμη το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το λειτουργικό κόστος και δεν μιλάω τώρα για τους διάφορους παράγοντες που είναι σε κόκκινο και σε μπλε όπως βλέπετε στη διαφάνεια αλλά Βλέπετε ότι υπήρχε αύξηση το 2007, δηλαδή το 2007 ήταν κακή χρονιά για το σύνολο της κτηνοτροφίας ε, και της παραγωγής βοδινού κρέατος. Όταν βλέπουμε την εξέλιξη μεταξύ 2005 και 2008... Μόνο για το λειτουργικό κόστος βλέπουμε ότι η εξέλιξη ήταν πολύ έντονη. 9 με 38% αύξηση σε σχέση με το 2005 βέβαια αφορούσε κυρίως το σύστημα, τα συστήματα που, ε, που βασίζονται κυρίως στην αγορά ε, ζώων και όχι τόσο στην παραγωγή στη φάρμα. Όταν βλέπουμε λοιπόν το λειτουργικό κόστος εκτός ε, της ε, αγοράς, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση Δηλαδή ε, προσπάθησαν να ε, μειώσουν την παραγωγή για να μειώσουν και τον κόστος. Βλέπουμε τώρα πώς είναι το σύστημα του 2007. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη οι διαφορές ε, είναι πολύ μεγαλύτερες για την παραγωγή του ε, ε, βοδινού κρέατος σε σχέση με την πάχυνση. Βλέπουμε δηλαδή 1,5 μέχρι 3 ευρώ ανά κιλό ζώντος κρέατος, κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την κατάσταση που υπάρχει στην πάχυνση και Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι παράγοντες και σταθεροί, ε, όπως για παράδειγμα η οικογενειακή εργασία και η μισθωτή εργασία που συνυπολογίζονται. Ε, υπάρχει επίσης και άμεση εξάρτηση του τομέα από τις επιδοτήσεις ε, και επομένως ε, η αποσύνδεση ή μη είχε και αυτή το αποτέλεσμά τη σε σχέση για παράδειγμα με τις βιολογικές καλλιέργειες και την κατάσταση που βλέπουμε στην Γερμανία. Όταν δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, ε, και αυτά είναι αποτέλεσμα ενός ε, παγκόσμιου πάνελ, ε, του οποίου ηγείται ένα γερμανικό πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτό το πάνελ, το Agri Benchmark, μας δίνει κάποια αποτελέσματα. Το δεύτερο σύστημα είναι ένα ισπανικό σύστημα ε, και έχουμε επίσης και τρία άλλα συστήματα, το βραζιλιάνικο, το ε, αυστραλέζικο και το ε, καναδέζικο. Το κόστος παραγωγής στην Ιρλανδία και στην Ισπανία είναι συγκρίσιμο σε σχέση με τις τέσσερις χώρες που εξετάσαμε προηγουμένως, ενώ στη Βραζιλία και στον Καναδά το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο. Δηλαδή ο συντελεστής είναι 1 έως 3 όταν το συγκρίνουμε με την ευρωπαϊκή παραγωγή όχι μόνο λόγω του κόστους ε, των τροφίμων, των τροφών, αλλά και του κόστους παραγωγής, ε, του κόστους ε, της εργασίας που είναι επίσης πολύ χαμηλότερο. Στις τρίτες αυτές χώρες, και στη Βραζιλία και στον Καναδά, δεν έχει καλυφθεί το κόστος της παραγωγής, δεν έχει καλύψει το κόστος της παραγωγής, το κόστος ε, των ε, διαφόρων ε, συντελεστών. Υπήρξαν διάφορα, διάφορα σενάρια εξέλιξης, για παράδειγμα μια συμφωνία στον ΠΟΕ βάσει των όσων υπήρχαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο του 2008. Υπήρχε ένα σενάριο μείωσης επιδοτήσεων κατά 25% ε, μέχρι το 2013 και κάναμε σύγκριση για το βοδινό κρέας. Εκτιμάται ότι οι εσωτερικές τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 23%. Επομένως, το σύνολο των συστημάτων βασίζεται πάρα πολύ σε ένα σύστημα για παράδειγμα συμφωνίας με τον ΠΟΗ, ειδικότερα για ευαίσθητα προϊόντα που έχουν ε, συγκεκριμένες δασμολογικές, ε, συγκεκριμένα δασμολογικά ε, καθεστώτα. Και το ίδιο ισχύει και με την πάχυνση, γιατί εκεί ο τομέας πλήρεται πολύ περισσότερο. Βέβαια, το το, το σύστημα βασίστηκε... Ε, χωρίς να λάβουμε, βασιστήκαμε ε, στο, σύστημα αυτό χωρίς να λάβουμε υπόψη κάποιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ειδών κρέατος. Επίσης δεν λάβαμε υπόψη τόσο την αποσύνδεση, κάτι το οποίο ενδεχομένως περισσότερους κτηνοτρόφους να τους επηρέαζε περισσότερο από κάποιους άλλους. Ακόμη και αν δεν υπήρχε συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Οι ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι εξαρτώνται πάρα πολύ από τις τιμές των, τροφών, των ζωοτροφών ε, και δεν έχουν και ιδιαίτερα περιθώρια ε, ελιγμών. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο δεν ε, επιδέχεται ιδιαίτερη προσαρμογή. Σε σχέση με το ισπανικό σύστημα βέβαια μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες αγορές που μπορούν να πουλήσουν οι κτηνοτρόφοι τα προϊόντα τους ακριβότερα από ό,τι σε άλλες αγορές. Ε, τώρα μιλάμε για ε, πολύ συγκεκριμένα είδη κρέατος βέβαια, τα οποία μπορούν να πουλούνται ακριβότερα στην Ισπανία από ό,τι κάπου αλλού. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της παραγωγικότητας της ε, εργασίας, το οποίο συνυπολογίζεται σε κάποια συστήματα, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση των επιδοτήσεων, του συστήματος επιδοτήσεων. Να περάσουμε τώρα ε, στο πρόβιο κρέας ε, Έγινε λοιπόν μελέτη και για το συγκεκριμένο τομέα. Πρόκειται για τον τομέα που εδώ και 20 χρόνια αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα ζωικό κεφάλαιο το οποίο μειώθηκε κατά 1 πέμπτο εδώ και 18 χρόνια. Έχουμε μία μείωση ζωικού ε, κεφαλαίου το οποίο ειδικότερα ε, μειώθηκε ακόμη περισσότερο εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε μία μείωση της τάξεως του 4% για το ε, ζωικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης των Επίσης, έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ε, γιατί ούτως ή άλλως τα περισσότερα πρόβατα ε, εκτρέφονται στις ε, μειονεκτούσες περιοχές και αν δεν γίνεται αυτή η αν δεν υπάρχει αυτή η κτηνοτροφική δραστηριότητα, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στην περιοχή. κάτι το οποίο βέβαια έχει αμέσως σχέση και με το γαλακτοκομικό τομέα γιατί ε, στην Νότια Ευρώπη είναι πολύ συνδεδεμένο ο τομέα αυτός με το γάλα, στις βόρειες χώρες λιγότερο. Βέβαια στη Γαλλία η κατάσταση είναι κάπως ενδιάμεση. Επίσης, στηριχθήκαμε σε συστήματα με προορισμό το κρέας στην Ιρλανδία, στη Γαλλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαπιστώνουμε ότι το λειτουργικό κόστος στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για συστήματα ε, που βασίζονται κυρίως σε βοσκοτόπους ε, με γρασίδι, βλέπουμε ότι στην Γαλλία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπετε για παράδειγμα το το μπλε κομμάτι της διαφάνειας δεν έχει καμία σχέση στη Γαλλία ε, με τις υπόλοιπες χώρες και αυτό φαίνεται καθαρά. Με την εξαίρεση βέβαια του τελευταίου συστήματος, ε, του συστήματος ε, του, του κτηνοτροφικού, και βλέπουμε επίσης ότι ε, στη Γαλλία ε, το 40% καλύπτεται των αναγκών ε, του πρόβειου κρέατος με την τόπια, από την τόπια παραγωγή ενώ. Τώρα, όσον αφορά τον αντίκτυπο ειδικότερα του, κόστους, ε, του λειτουργικού κόστους στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται αυτό το ε, σύστημα ε, των, ε, των βοσκοτόπων υπήρξε και μεγαλύτερη αντίσταση στην κρίση που αντιμετώπισε ο τομέας. Τώρα, στη Γαλλία υπήρξε μία απόφαση να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο ε, τα ε, πουλερικά, κάτι το οποίο βέβαια ανακουφίζει κατά κάποιο τρόπο τον τομέα, στη Γαλλία τουλάχιστον. Ειδικότερα αν μειωθούν οι επιδοτήσεις ε, κατά 25% μετά το 2013, το σύστημα στη Γαλλία τουλάχιστον θα, θα πληγεί πάρα πολύ στις υπόλοιπε χώρε μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο ο αντίκτυπο, αλλά παρόλα αυτά θα υπήρχαν κάποιες συνέπειε. Ειδικότερα λοιπόν όλες ε, οι χώρες που βασίζονται σε αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην αύξηση του κόστους, αλλά βέβαια υπάρχουν και μεγάλες ανισότητες ε, στο εισόδημα από τις δραστηριότητε αυτέ. Ε, και επίσης πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες αύξησης της παραγωγικότητας εργασίας τους προς αυτό. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα, ειδικότερα στην περίπτωση των... Ε, ε, Θα δώσω τώρα το ε, λόγο στον συνάδελφο να σας μιλήσει για τα πουλερικά. Για τα πουλερικά. Μπορεί, να είναι, μιλάω για παραγωγή κρέατος, για κατανάλωση από πουλερικά, πάπιες και άλλα συναφή, όρνηθες και αυτά. Η βασική παραγωγή είναι ε, χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και δεν υπάρχουν ε, μεγάλες ε, διαφορές ε, στην παραγωγή τους ε, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία είναι επίσης σημαντικές χώρες παραγωγής και αλλά έχουν πολύ χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές είναι οι τρίτες χώρες, 30 με 40% χαμηλότερο κόστος παραγωγής στη Βραζιλία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό βέβαια είναι το κόστος παραγωγής στο επίπεδο μονάδας, φάρμας. Ε, και μπορεί η διαφορά αυτή της ε, τιμής παραγωγής να διευρυνθεί πολύ περισσότερο. Οι χώρες αυτές χαμηλού κόστους παραγωγής όπως η Βραζιλία ε, παράγουν και τις ζωοτροφές, ε, τη σόγια, ε, καλό κλίμα, καλές συνθήκες. Έχουν λοιπόν πολύ εύκολη πρόσβαση στις ζωοτροφές, χαμηλό κόστος εργασίας και πολύ λιγότερες κανον, ρυθμίσεις, κανονισμούς, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο δηλαδή όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων από ότι στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς λόγω όλων αυτών των παραμέτρων η παραγωγή του είναι πολύ φθηνότερη από την Ευρώπη ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τώρα τα εισοδήματα στην Ολλανδία και στη Γαλλία. Οι χώρες αυτές ε, έχουν μια πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά την παραγωγή. Η Γαλλία έχει ένα ε, ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ε, συμβάσεις ε, παραγωγής με τους διάφορους παραγωγούς ενώ η Ολλανδία και η Πολωνία δεν έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα με συμβάσεις, ειδικά συμβόλαια παραγωγής. Το 2008 είναι, ήταν μια χρονιά πολύ, πολύ χαμηλών εισοδημάτων ε, βλέπετε όμως ότι η Γαλλία είχε ένα πολύ, πολύ σταθερότερη πορεία, η οριζόντια κόκκινη γραμμή, ενώ η Ολλανδία είχε πολλά ανεβοκατεβάσματα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν οι δύο χώρες αυτές, Ολλανδία και Γαλλία, είχαν χαμηλά εισοδήματα η παραγωγή. Τώρα όσον αφορά την, ε, τον ανταγωνισμό, τη Βραζιλία το κατεψυγμένο φιλέτο, κατεψυγμένο φιλέτο στήθος πουλερικών και αυτά τα κομμάτια η Βραζιλία μπορεί να τα προσφέρει στην Ευρώπη στη μισή τιμή. Ε, με το μπλε βλέπετε εδώ είναι τα, οι πολύ υψηλή εισαγωγική δασμοί που πρέπει να καταβληθούν για την εισαγωγή στη Βραζιλία αυτού του κατεψυγμένου κρέατος αλλά ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός γιατί προσφέρονται σε χαμηλή τιμή δεν υπάρχει σύστημα ποσοστώσεων, αλλά ακόμα και χωρίς ποσοστώσεις και με την καταβολή πολύ υψηλών δασμών εισαγωγής, ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός με την Βραζιλία. Είναι λοιπόν σαφές από το διάγραμμα αυτό ότι υπάρχει μία ανισορροπία ε, στις εμπορικές συναλλαγές. Καταλήγοντας τώρα με, το, με την παραγωγή. Εδώ βλέπετε τα δια... σύγκριση, συγκριτικό πίνακα διαφόρων συστημάτων παραγωγής, ολοκληρωμένο σύστημα, μη ολοκληρωμένο. Το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ε, παρουσιάζει μια καλύτερη σταθερότητα εισοδημάτων για τους παραγωγούς και μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στα διάφορα, στην αλλαγή των σημάτων που δίνει η αγορά και μπορεί να προσαρμοστεί και σε καινοτομίες τα μη ολοκληρωμένα συστήματα, Ολλανδία, Πολωνία, εδώ η παραγωγή είναι πιο καινοτόμοι, ενεργούν πιο επιχειρηματικά, αλλά μπορούν να αντιδράσουν με πολύ αργότερους ρυθμούς. Τώρα, η, τα, τα πουλερικά προς ε, κατανάλωση κρέας πουλερικών. Εδώ βλέπουμε Ολλανδία, Πολωνία, Γαλλία, χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερες τιμές που πληρώνονται για το κρέας, αλλά το, ε, πρέπει να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό που είναι πολύ ε, σκληρός. Και τώρα το υψηλό επίπεδο η υψηλή η υψηλή ποιότητα, το η κόκκινη ετικέτα από τη Γαλλία έχει πολύ ψηλότερο κόστος παραγωγής, σχεδόν το διπλό, αλλά περιορισμένη αγορά διάθεσης, ε, ε, διότι είναι πολύ ακριβά τα προϊόντα αυτά, έχουν όμως τη βούλα της ανώτερης ποιότητας. Υπάρχουν λοιπόν προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται στην Ευρώπη. Ε, όσον αφορά τώρα τα χειροτροφία, εδώ βλέπετε στα αριστερά το κόστος παραγωγής στις βασικές χώρες Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία. Ε, τα ίδια συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε και για το βόλιο κρέας, όπως εδώ για το χείριο. Ε, ίδια διακύμαση του κόστους παραγωγής, λίγες οι διαφορές. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ε, στον πίνακα αυτό, θα μπορούσαμε δηλαδή και τη Δανία και στα δεξιά βλέπετε πάλι το κόστος παραγωγής ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία περίπου 60-40% χαμηλότερο κόστος και πάλι λόγω των ιδίων ε, παραγόντων που επικρατούν ε, φτηνή και γρήγορη πρόσβαση σε ζωοτροφές, φτηνό εργατικό κόστος κλπ. Ε, τώρα τα οικογενειακά εισοδήματα στη χειροτροφία. Ε, εδώ έχω συγκριτικού πίνακες Ολλανδίας και Γαλλίας. Βλέπετε τον, τις διακοιμάνσεις των εισοδημάτων ε, προς τα άνω φθήνους, προς τα κάτω, πάνω κάτω, πολύ μεγάλες διαφορές. Τη μία χρονιά πολύ καλή κατάσταση εισοδημάτων, την άλλη λίγα αρνητική. Είναι λοιπόν σαφής αυτή η αστασής πορεία των εισοδομάτων. Ε, το άμεσο, το, ε, ο μέσος όρος είναι 25 με 30.000 ευρώ το χρόνο, το μέσο εισοδήματος μονάδα δηλαδή, αλλά με μεγάλες διακοιμάνσεις από χρόνο σε χρόνο. Ε, σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε τα εισοδήματα κατά ε, αναέτος στη Γαλλία και στην Ολλανδία υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από ε, μονάδα σε μονάδα. Δεν υπάρχει μέσος όρος που μπορούμε να αναφερθούμε. Ορισμένες φάρμες έχουν πολύ καλή πορεία, άλλες όχι και βλέπετε την πολύ μεγάλη διακύμανση των εισοδημάτων μεταξύ των παραγωγικών μονάδων. Εξαρτάται αυτό και από την δίκευση που έχουν στα προϊόντα που παράγουν. Και καταλήγοντας με τον διεθνή ανταγωνισμό, βλέπετε όπως και με την, ε, τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής έχουμε μια ειδική, ειδικά έντονη, έντονο ανταγωνισμό τη Βραζιλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε για το στήθος και τα φιλέτα κοτόπουλου ε, ε, ε, αριστερά βλέπετε το κομμάτια όχι στήθος, όμου Ε, εδώ πληρώνονται υψηλοί δασμοί ε, εισαγωγής. Αν οι δασμοί αυτοί μειωθούν, τότε θα δημιουργηθεί μεγάλη διστρέβλωση του ανταγωνισμού. Προς το παρόν ο ανταγωνισμός κρατιέται σε κάποια όρια επειδή είναι υψηλοί οι δασμοί ε, εισαγωγής. Παραγωγή, χειροτροφία και διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εδώ στην Ολλανδία και στη Δανία έχουμε πάρα πολύ καλές φάρμες, πολύ καλές μονάδες που ε, ειδικεύονται με υψηλά εισοδήματα αλλά μεγάλες διακοιμάνσεις ανά έτος. Ε, άλλες ειδικευμένες μονάδες στην Ολλανδία, Δανία και Γαλλία, ολοκληρωμένες μονάδες ε, χαμηλότερα εισοδήματα, ε, κίνδυνοι μεγάλα ρίσκα που αναλαμβάνουν και λιγότερες διακοιμάσεις εισοδήματος. Μεσαίες μονάδες χειροτροφικές, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλό ρίσκο και αποζημιώσεις ε, ε αποζημιώνονται για τα χαμηλά εισοδήματα με άλλες δραστηριότητες, παραδείγματο χάρη, παραγωγή γάλακτος και καλλιέργειας δημητριακών και έχουμε και μικρές φάρμες ε, χειροτροφικές, Πολωνία και Γερμανία που έχουν χαμηλότερη απόδοση, υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά είναι πιο ευέλικτες. Αυτά, ευχαριστώ. Το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης αφορά στις συστάσεις. Είναι ε, κάτι το οποίο έχουν επεξεργαστεί οι διάφοροι εμπειρογνώμονες και αυτό το ερωτηματολόγιο έχει προβλεφθεί σε 55 συμμετέχοντες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε άλλες χώρες. Οι συστάσεις αυτές λοιπόν είναι χωρισμένες σε 5 κεφάλαια. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες από τη σελίδα 17 από 17 μέχρι 22 της έκθεσης ε, δεν βρίσκονται στο, στην περίληψη. Το πρώτο κεφάλαιο το είδατε πολύ καλά διότι εκεί αναφέραμε την, ε, την όλη παρουσίασή μας, το θέμα της, ε, του διεθνούς ανταγωνισμού. Μία συμφωνία στον ΠΟΕ θα επηρέαζε πολλούς ε, αγροτικούς τομείς, αλλά ιδιαίτερα τον τομέα του κρέατος στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν μετά από πολλές συζητήσεις συστήνουμε να περιορίσουμε δραστικά την μείωση των δασμών για τα προϊόντα, για τους, φόρους, για τους δασμούς και τους φόρους που αφορούν τα ευαίσθητα προϊόντα. Και προτείνουμε λοιπόν μια χρονική περίοδο προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία του ΕΕ. Μιλήσαμε επίσης για σύμμετρες ε, κανόνες. Ε, ακούσατε στο πρώτο τμήμα του πρωινού αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κανόνες που είναι πολύ πιο αυστηροί στην Ευρώπη από ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου και πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα χρονοδιαπραγμάτευση και στον ΠΟΕ και στο Κόδεξ Αλιμεντάριου αλλά και στο Γραφείο Επιζωτιών. Μου ζητούν να βιαστώ, γι' αυτό θα μιλήσω πιο γρήγορα. Αλλά όλα αυτά φυσικά οδηγούν σε υπερβολικό κόστος, σε αύξηση του κόστους τη τάξη του 5-10% σύμφωνα με τα συστήματα και με τους τομείς, με τους Μιλάμε πολύ για το ζήτημα της υγείας ε, των καταναλωτών αλλά και των ζώων αφορούν τις τομείς ε, της καλής μεταχείρισης, περιβαλλοντικούς ε, κλπ. Προτείνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει πολλά περισσότερα σε ό,τι την παρουσία της στους διεθνούς οργανισμούς, αλλά και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσει να μην είναι και πολύ μπροστά, να μην ηγηθεί Εκτό εάν θέλει να προωθήσει μέτρα που αφορούν προστασία του περιβάλλοντος ή την προστασία των ζώων, την καλή μεταχείρισή του κλπ. Μιλάμε, προτείνουμε μάλλον την γενίκευση του σήμανση ε, σχετικά με τη χώρα καταγωγή πρόελευση, διότι αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο στο πνεύμα του καταναλωτή με του κανόνε που ισχύουν και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στι χώρε αυτέ. Βλέπουμε λοιπόν πω ο διεθνή ανταγωνισμό γίνεται προϊόν που είναι διαφορετικά όπως το αλατισμένο κοτόπουλο ή το βόλιο κρέας το οποίο μπορεί να πωλείται ως φρέσκο αλλά στην ουσία είναι κατεψυγμένο για τρεις-τεσσέρις μήνες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο κανονής να γνωρίζει τι αγοράζει. Δεύτερον, ε, ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικές ε, ανησυχίες, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε απαντού, πανταχού, ειδικά σε ό,τι φορά την ε, αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, μια τυποποίηση της, του υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό να ενταθούν οι έρευνε για τη μείωση των εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, να στήσουν τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια για, και να προωθήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της ενώσεων πηγών ενέργειας, ε, αιωλική, υδραυλική κλπ. Και επίσης θα πρέπει να παροτρύνουμε αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά benchmarking, δηλαδή ομάδα προβληματισμού και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο εκτροφέων στην έκθεση θα παρατηρήσετε πως ε, μια, ένας από βασικούς λόγους για την έκρηξη των τιμών στα τρόφιμα είναι η πολιτική επί των καυσίμων και όταν ε, παροτρύνουμε την αύξηση τη τιμή ενός ε, καυσίμου, ταυτόχρονα αυξάνουμε και τις ε, τιμές, το, το κόστος μάλλον του παραγωγού. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα προϊόν το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκτροφής, από εκτροφής κλπ. για το οποίο θα οδηγούσε μια μείωση ενδεχόμενα του κόστους παραγωγής. Τρίτο κεφάλαιο, πώς να αντιμετωπίσουμε την πτυτικότητα των τιμών, τις διακυμάνσεις που είναι κάτι το οποίο πρέπει να νομίσουμε τα επόμενα 5-10 χρόνια. Υπάρχουν προτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρουμε πως ε, η εκμετάλλευση είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην αύξηση των τιμών. Αυτό μπορεί να Γι' αυτό οδηγεί σε προβλήματα στις ε, πιο φτωχές χώρες. Αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το ΙΦΑΟ. Ξέρουμε πως η κερδοσκοπία επηρέασε σημαντικά την αύξηση των τιμών των δημητριακών και των σπόρων και κάποια μέσα ρύθμισης των αγορών που έχουν απομείνει μετά από τον διαγνωστικό έλεγχο της ΚΑΠ θα πρέπει να διατηρηθούν όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση αλλά και κάτι το διαφυσβητούμενο όπως οι επιστροφές. Εμείς βλέπουμε με χρησιμότητα των επιστροφών σε περίπτωση σοβαρής κρίσης σε ό,τι αφορά τις συναλλαγματικές οτιμίες. Αυτές αποτελούν ένα όπλο το οποίο είναι διάφανο θα έπρεπε λοιπόν να μπορέσουμε στην Ευρώπη να αντιδράσουμε με τις επιστροφές σε αυτές τις ε, συναλλαγματικέ οτιμίες και διακοιμάσεις τους. Στην έκθεση θα βρείτε διάφορα στοιχεία αναφορικά με το καναδικό σύστημα που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ζητήσουμε την ε, σύνδεση για σε φορά την πλημοδότηση της ε, δασοφόρας Αγελάδας ε, και μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανία κρέατος ε, έχει ανάγκη από στήριξη, από το κεφάλαιο, πως ε, να περιορίσουμε το υπερβολικό κόστος που άπτεται των προτύπων και της υπερβολικής, των υπερβολικών ρυθμίσεων. Για κάθε νέο κανονισμό που θα επηρέαζε το κόστος παραγωγής και σκέφτομαι εδώ το θέμα της μεταφοράς ζών των ζών, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώσουμε διότι έχουμε ξεπεράσει το ωράριο των διερμηνέων. Λοιπόν, τα όσα απομένουν θα τα διαβάζετε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λυπάμαι που έχω